σας. Υποθέτω, φαντάζομαι ότι δεν είναι και η τελευταία φορά που συζητάτε για τη συμφωνία αυτή με τη Μερκοσούρ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πιστεύω ότι δεν θα είναι η τελευταία φορά, κύριε Επίτροπε. Προς το παρόν όμως κλείνει η συζήτηση, κοινή συζήτηση για τη Μερκοσούρ. Και προχωρούμε στο επόμενο θέμα μας, στην αμερίστη διάταξη, που είναι η έκθεση του Αλάν Καντέκ, καθεστώς εισαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Προϊόντων Αλία και Ιδατοκαλλιεργία με προοπτική τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλλιευτική πολιτική και δίνω το λόγο ευθύ αμέσω στον κύριο Κατέρη. Τον εισηγητή για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, μια από τις βασικές ιδέες αυτής της έκθεσης είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια συνέπεια απαιτούμενη μεταξύ της ε, κοινή πολιτικής αλίας και της διεθνού μα πολιτική. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας που σήμερα βλέπουμε ότι η Επίτροπος Αλίας, η κυρία Δαμανάκη, βρίσκεται στα έδρανα της Επιτροπής. Είναι μια διαρκή μα συνομιλήτρια και ο Επίτροπος που είναι των με τα θέματα εμπορίου, ο κύριος Δεκούχτ. Είναι μεγάλη μα τιμή. Επιτρέψτε μου ωστόσο να θεωρήσω ότι αυτή η διπλή παρουσία από πλευρά επιτροπή εκτό από κολακευτική, είναι και αρκετά συνήθιστη. Για να δούμε τώρα την ίδια την έκθεση. Οι εισαγωγέ αλληλευτικών προϊόντων και προϊόντων καλλιέργεια από τρίτε χώρε προσωπούν το 60% τη κοινοτική κατανάλωση. Αυτό το επίπεδο εξάρτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ιδιαίτερα ενισχυτικό σε σχέση με τι εισαγωγέ, και είναι και αποτέλεσμα δύο αιτίων. Πρώτα απ' όλα τη ε, ελληπού κοινοτική παραγωγή και έπειτα γιατί όλο ένα και μεγαλώνει το άνοιγμα τη αγορά μα στι εισαγωγέ, λόγω των εμπορικών πολιτικών που σχεδιάζει η Επιτροπή εδώ και 10 χρόνια. Οι εξελίξει αυτέ λοιπόν δυσχεραίνουν ε, του ε, παραγωγεί αλίας τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν δυσκολίες με τιμές αρκετά υψηλές, ενώ η προσφορά είναι μικρότερη από τη ζήτηση σε πολλές περιπτώσεις. Οι προδιαγραφέ υγειονομικέ, περιβαλλοντικέ και κοινωνικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ψηλέ. Και με πικρία διαπιστώνουμε ότι οι ίδιε προδιαγραφέ δεν ισχύουν για τα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτε χώρε. Αυτό που διακυβεύεται λοιπόν εδώ είναι απλώς όχι μόνο η επιβίωση ενός ευρωπαϊκού τομέα παραγωγής ε, για μια οικονομικά εφόρο αλία, για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων, προϊόντων ποιότητας για τους καταναλωτές, αλλά και το θέμα της ε, πολιτιστικής διάστασης των παράκτιων περιοχών μας. Δεν είναι κάτι που μπορεί να διαπραγματευτούμε, κύριε Επίτροπε, η γαλλιευτική μας πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσουμε μια δασμολογική πολιτική σταθερή για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργεια και αλεία. Και η προτίμηση που δίδεται σε κάποιε τρίτε χώρε, ιδίω στι αναπτυσσόμενε χώρε, να ελέγχεται. Καθώ και να παρακολουθούμε του μηχανισμού του ΠΟΕ για να μπορεί να καλύπτουν οι ανάγκε ε, του μεταπητικού μα κλάδου. Δεν μπορούμε εδώ να ε, εφαρμόζουμε την ελβετική φόρμουλα ε, χωρίς διακρίσεις για ευαίσθητα προϊόντα. Επίσης, οι εμπορικές προτιμήσεις που δίνονται σε κάποιες τρίτες χώρες ε, θα πρέπει να σέβονται και τους υγειονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς ε, κανόνες που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ Και επίσης, η κύρια ευθύνη θα πρέπει να μετατοπιστεί από τι εμπορικέ διαπραγματεύσει για τα προϊόντα αλλία και υδατοκαλλιέργεια από τον Επίτροπο Εμπορίου προ τον Επίτροπο που είναι υπεύθυνο για τα αλληλευτικά προϊόντα και τι ναυτιλιακέ υποθέσει. Έτσι θα λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι ιδιαίτερε ανάγκε των προϊόντων αλλία και υδατοκαλλιέργεια. Ο... Αυτή η συζήτηση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και επί τη ουσία. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώ θα γίνει με την κοινή αλληλευτική πολιτική και επίση θα δουν, βλέπουμε ότι υπάρχει ατελμάτωση των διαπραγματεύσεων του κ. Δόχα στον ΠΟΕ. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει υπόψη να επαρκώ τι ανάγκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έπειτα, με την παρουσία του Επιτρόπου Ντεκούχτ, ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβλέψει δημόσιε διαβουλεύσει ώστε να σχεδιαστούν νέε κατευθυντήριε γραμμέ για την κοινή εμπορική πολιτική στα πλαίσια τη στρατηγική του 2020. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι πλέον ε, υπεύθυνο, είναι υπεύθυνο με τη διαδικασία τη συναπόφαση και για τα εμπορικά θέματα και για την εμπορική και την πολιτική αλεία. Θα πρέπει λοιπόν να κάνει τη φωνή του να ακουστεί και για τα ζητήματα αυτά. Και θα πρέπει να λάβουν υπόψη η Επιτροπή και το Συμβούλιο τι συστάσει που περιέχει η έκθεση αυτή. Σε κάθε περίπτωση θα επαγρυπνούμε του ερχόμενου μήνε και εγώ προσωπικά πρέπει να πω ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι για αυτό το σημαντικότατο ζήτημα. Σα ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Καρέ. Καλώ όριζα και την Επίτροπο κυρία Δαμανάκη και τη δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Καντέ και τις ε, επιτροπές του Κοινοβουλίου που ε, ανέλαβαν αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας εκφράσατε τη λύπη σας για το ότι η πράσινη βίβλος για την κοινή αλληλευτική πολιτική δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τα ζητήματα που ανακοινώσατε εδώ. Και εγώ σας το έχω σήμερα εδώ. Έχω να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή είναι ε, αποφασισμένη εργαστή λαμβανωμένων υπόψη όλων των πολιτικών που επηρεάζουν τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Όπω είπα και νωρίτερα, στόχο πολιτική είναι να ανατρέψει την αρνητική το φαύλο κύκλο μέσα στον οποίο βρισκόμαστε τώρα. Έχουμε έναν τομέα αλίας ούτε οικονομικά βιώσιμο, ούτε και ε, τεχνολογικά βιώσιμο. Χρειαζόμαστε ισχυρή αλία με αξιοποίηση σωστή και εφόρο των πόρων, επιτρέποντας ταυτόχρονα και στον αλία την οικογένειά του και την κοινότητά του να ε, εξασφαλίσουν τα προστοζήν από τη δραστηριότητα αυτή. Χρειαζόμαστε λοιπόν και την ικανοποίηση των αναγκών των αγορών των εσωτερικών και των διεθνών, αλλά και τώρα και για το μέλλον. Και βεβαίως ακούω τις ε, διαμαρτυρίες σας για, ε, για τον αθέμητο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες, για τις συνθήκες ε, τις κοινωνικές, τις περιβαλλοντικές που δεν τηρούνται την νομοθεσία για την προστασία της υγείας. Σας διαβεβαιώ ότι την ίδια αυτή ανησυχία εξέφρασαν και όλα τα κράτη-μέλη που μίλησαν στο τελευταίο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας. Άρα πρέπει εδώ να δοθούν απαντήσεις. Και ενώ ε, αναθεωρούμε τους κανόνες για την κοινή αλληλευτική πολιτική στο πλαίσιο της μεταρρυθμίσης αυτής, μια από τις μεγαλύτερες μας προκλήσεις θα είναι να εξασφαλίσουμε ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για όλα τα προϊόντα που θα μπαίνουν σε ευρωπαϊκές αγορές. Ως εκ τούτου και εν προκειμένου πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί για την σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας, ώστε να αποτραπεί η αρρύθμιστη, η παράνομη και η μη δηλωμένη αλληλεία. Επίσης, πρέπει να ε, ε, επαγρυπνούμε ώστε να τηρούνται όλοι οι διεθνείς κανόνες και από τους εταίρους μας και να φροντίζουμε να παρακολουθούμε αν τηρούν με σοβαρότητα τους κανόνες τους, της βαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής προστασίας. Βεβαίως και ακούω τις εκκλήσεις για τήρηση αυστηρή και συνεπή των πολιτικών μας. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη και ευρεία πολιτική. Δύο τρίτα των ε, ψαριών που καταναλώνονται στην Ευρώπη εισάγονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται για τη μεταποιητική μας διαδικασία σταθερή ροή προϊόντος και σταθερή τιμή για τον καταναλωτή. Ένα τρίτο της αγοράς πάντως καλύπτεται από τον ευρωπαϊκό κλάδο που εξασφαλίζει και τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας και έτσι διαφυλάσσει τον κοινωνικό ιστό σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Και έτσι, ενώ βρισκόμαστε σε ένα ε, στο πλαίσιο μιας μεγάλης αναθεώρησης κοινής αλληλευτικής μας πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται και να λάβει υπόψη το περίπλοκο χαρακτήρα του κλάδου της αλίας, αλλά και τις οικονομικές πραγματικότητες και τα οικονομικά δεδομένα. Εγώ προσβλέπω σε πολύ καλή συνεργασία με τον συνάδελφο κύριο Ντεγκιούχτ, έτσι ώστε να προσδιορίσουμε εγκαίρως και να δώσουμε επαρκές χρονικό περιθώριο για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να προχωρήσουμε σωστά στη μεταρρύθμιση αυτή τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Για δε τι διαπραγματεύσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε και με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούμε τι συστήσει περί επιδοτήσεων, γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πάντοτε σε θέση να υποστηρίζουμε περιβαλλοντικά μέτρα και πρωτοβουλίε των κρατών μελών. Για δε την αναθεώρηση της ε, πολιτικής σχετικής με την αγορά, συμφωνώ με το σχέδιο της έκθεσης στο ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν τα μέσα της κοινή οργάνωσης αγοράς και η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει να ενισχύσει τις οργανώσεις των παραγωγών και τη δυνατότητά τους να συνδυάζουν καλύτερα, να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αλυσίδα της ζήτηση και της αγοράς με τα προϊόντα τους. Ταυτόχρονα πρέπει να επιδιώξουμε σταθερότητα στην αγορά και στην προσφορά και ενημερώσει και ικανοποιητική ε, πληροφόρηση του καταναλωτή, δηλαδή σήμανση. Γιατί ο καταναλωτής θέλει να γνωρίζει περισσότερα για το προϊόν που αγοράζει, θέλει να γνωρίζει πού ε, πιάστηκε το ψάρι ή που ήταν η χθεοκαλλιέργεια, εάν τηρήθηκαν οι κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας και η αηφόρος αλία. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τεθειμένη να τηρήσει αυτές τις προδιαγραφές και να προσφέρει με τους κανόνες που θα ορίσει την επαρκή ενημέρωση των καταναλωτών. Για δε την ηχθειοκαλλιέργεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στρατευμένη στην τήρηση των κανόνων για μια αηφόρο ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών, όπως έχουμε συζητήσει άλλωστε και μέσα από τη σχετική έκθεση. Και επίσης συμφωνούμε ότι η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυσσόμενη μπορεί να περιορίσει την εξάρτησή μας από τις εξαγωγές και να, δώσει περισσότερη, να ικανοποιήσει περισσότερο την αναπτυσσόμενη ε, ζήτηση στα αλληλευτικά προϊόντα. Και κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι προσβλέπουμε σε μια πολύ σημαντική συμβολή από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη μεταρρύθμιση τη κοινή ελευθερική πολιτική και ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει ένα πολύ σαφέ πολιτικό μήνυμα για όλου του ε, και τι αλληλεί μα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνουν μια πολύ σκληρή δουλειά και ταυτόχρονα περιμένουν σε αυτό το μήνυμα για το μέλλον του. Ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο. Ο κύριο Δεχούχτ, παρακαλώ να μα δώσει τι του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Η Επιτροπή ευχαριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απόφασή του να αναλάβει έκθεση πρωτοβουλία όσον αφορά τα προϊόντα αλίας. Η συζήτηση αυτή στο Κοινοβούλιο μας βοηθάει να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις που κάνουμε όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Καλό τους ευρωβουλευτές να λάβουν υπόψη τους τις εξή παρατηρήσεις όσον αφορά τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή γνωρίζει τη φύση του ελευθερικού τομέα. Γνωρίζει πόσο σημαντικός είναι αυτός για ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινότητα και αυτό λαμβάνεται υπόψη στην εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σας πω ότι πρέπει να συμφιλιώνουμε πολλά και διαφορετικά συμφέροντα όλων των πλευρών που εμπλέκονται στον αλληλευτικό τομέα. Είτε πρόκειται για τους παραγωγούς, είτε πρόκειται για τους μεταπητές, είτε πρόκειται για τους καταναλωτές. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να συνεχίσει την πολιτική της για τα αλληλευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και να έχει μια ισορροπημένη λύση όσον αφορά την προμήθεια τέτοιων προϊόντων που να συνάδει με την ζήτηση που έχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προστατεύοντας πάντα τους στόχους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαρτώμενη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά προϊόντα αλίας και υδατοκαλλιέργειας για να ικανοποιήσει τη ζήτηση στην αγορά της. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη ζήτηση των καταναλωτών, αλλά και με τις τάσεις που υπάρχουν, με την εξάρτηση που υπάρχει. Γι' αυτό και η μεταρρύθμιση της κοινή ελευθερικής πολιτικής είναι μια καλή ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ενισχύσει την απόδοση του τομέα και να γίνει αυτός πιο ανταγωνιστικός παγκοσμίω. Οι τάσεις θα συνεχιστούν. Το ξέρουμε αυτό και σε πολυμερές επίπεδο και σε διμερές επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο θα συνεχιστούν οι ίδιες οι τάσεις. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν και λαμβάνει υπόψη της και έχει λάβει υπόψη της και θα λαμβάνει υπόψη της την κατάσταση στις αγορές και θα φροντίσει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων που υπάρχουν όπως σας είπα και πριν. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των τάσεων που έχουμε σε διεθνές επίπεδο θα κάνουμε τις προσαρμογές που χρειάζεται, λαμβάνοντας υπόψη μας το ρυθμό της μεταρρύθμισης της κοινή ελληνικής πολιτικής. Θα αναφερθώ τώρα σε μία από τις κύριες προτάσεις που αναφέρονται στην έκθεση και που είναι η δυνατότητα ε, προϊόντων ε, αλληλευτικών νάμα. Σε αυτό το πλαίσιο των συζητήσεων υπάρχει μεγάλη δυσκολία να ξεχωρίσουμε τα αλληλευτικά προϊόντα από τα νάμα. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα παρά την μεγάλη πίεση που αντιμετωπίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει τα όσα αναφέρει η εκθεσή σα για τις δυνατότητες διαπραγματεύσεων που υπάρχουν όσον αφορά τα προϊόντα αυτά, ώστε να περάσουν από το εμπόριο στην αλία. Όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντως είναι συνολικά υπεύθυνα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι και ο Επίτροπος Εμπορίου είναι υπεύθυνος για τις διαπραγματεύσεις αλλιευτικών προϊόντων. Δεν δρούμε μόνοι μας, αλλά συλλογικά διαπραγματευόμαστε σε συνεργασία με ε, ε, την ε, Γενική Διεύθυνση για την Πολιτική στη Θάλασσα, για παράδειγμα. Η Επιτροπή θέλει να διαβεβαιώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίε σα όσον αφορά τον αληφτικό τομέα στι διαπραγματεύσει. Η Επιτροπή στηρίζει τα συμφέροντα του τομέα τη Ευρωπαϊκή Ένωση στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και λαμβάνουμε υπόψη μας και τις ευαισθησίες που υπάρχουν παρόλο που δεχόμαστε τεράστιες πιέσεις από τους εμπορικούς μας εταίρους. Θέλουμε να στηρίξουμε τα συμφέροντα λοιπόν των Ευρωπαίων Αλλιών και προσπαθούμε να άρουμε ό,τι εμπόδια υπάρχουν ακόμα και που θέτουν οι εμπορικοί μας εταίροι όσον αφορά τις εξαγωγές της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έτσι ώστε ακριβώ να υπάρχει ισορροπία και ισοτιμία στις σχέσεις μας. Τέλος, η έκθεση ζητάει ισοτιμία όσον αφορά τα αλληλευτικά μας προϊόντα σε σχέση με τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προωθήσει υψηλού επίπεδου ε, προϋποθέσεις ποιότητας για να ανοίξει τις αγορές της. Και αυτό συμπεριλαμβάνεται στις εμπορικές μας συμφωνίες και σε διάφορα διεθνή φόρα. Το λέμε αυτό. Στα Ηνωμένα Έθνη, στο ΦΑΟ και σε περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλληλευτικών προϊόντων. Το λέμε και το ξαναλέμε και επαναλαμβάνω. Θέλουμε και είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να συνεχίσουμε να συζητάμε με τους ευρωβουλευτές για τις διαπραγματεύσεις τις εμπορικέ που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά προϊόντα αλίας και υδατοκαλλιέργειας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαντόχη τώρα το λόγο για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, νομίζω εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει σύγκληση της Επιτροπής Αλίας και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου. Ε, και σε αυτό, σε σχέση, αυτό σε σχέση με τη διαπίστωση και τις προτάσεις μας ε, σε αυτό το πλαίσιο. Ε, υπόθηκε ήδη η αλία είναι ένα τομέα σημαντικότατος και για την χωροταξία και για την πολιτιστική ταυτότητα και για την απασχόληση και στην Ευρώπη. Είναι ένας τομέας ο οποίος σήμερα δεν είναι αρκετά ισχυρός ε, λόγω των αποθευτικών αλλιευμάτων όπως έχουν διαμορφωθεί. Υπάρχουν πάρα πολλά αποθέματα σήμερα τα οποία τα υπερεκμεταλλευόμαστε. Επίσης σήμερα την να μας που νοήσουν ότι ο στόχο τη κοινή αλληλευτική ε, πολιτική τη Ευρώπη θα πρέπει να είναι η προσαρμογή μα ε, στην παγκοσμιοποίηση την εμπορική. Αυτό έχει ένα πολύ σοβαρό αντίκτυπο στην αλία και από κοινωνική και από οικονομική άποψη, αλλά και από περιβαλλοντική. Έτσι λοιπόν εμεί υπερασπιζόμαστε θερμά την ενσωμάτωση των κοινωνικών περιβαλλοντικών κριτηρίων στις εμπορικές συμφωνίες όταν μιλάμε για αλληλευτικά προϊόντα και στηρίζουμε την ιδέα ότι θα πρέπει να ε, αποσύρουμε, να βγάλουμε την αλία από τους τομείς νάμα των, ε, μη γεωργικών προϊόντων και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για θέματα επιστημιστικής ασφάλειας και βιοπικιλότητας. Από τη στιγμή όμω που θα τεθεί αυτό το θέμα στι διεθνεί μα διαπραγματεύσει, θα πρέπει η ευρωπαϊκή πολιτική να είναι υποδειγματική. Ε, να έχουμε περισσότερου αλληλεί που να αμείβονται καλύτερα και να μην, εκείνοι να μην υπεραλλιεύουν στα δικά μα ύδατα τα ε, αλλιεύματα, ούτε στα ύδατα στα οποία έχουμε αγοράσει δικαιώματα αλληλευτικά. Ευχαριστούμε. Και τώρα οι αγορητέ από τι πολιτικέ ομάδε, από το ΕΛΚΟ, κύριο Σαντινόρο, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπη, συνάδελφοι, ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Καντέκ για το έργο του, το οποίο ήταν εξαιρετικό για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως ε, το καθεστώς εισαγωγών ε, της Ευρώπης για τα ελληνικά προϊόντα. Όπως ετοίμαζα την παρέμβασή μου, σκεφτόμουν το θέμα της προσοχής που θα πρέπει να δοθεί στις εισαγωγές, ώστε τα εισαγόμενα προϊόντα να σέβονται τις ίδιες προδιαγραφές τις υγειονομικές Όμω σκέφτηκα ότι θα τα πούν άλλοι. Και επειδή δεν υπάρχει αρκετό χρόνο, θα παραμείνω στα εξή. Κάτι που θεωρώ ουσιώδε. Και κάτι που νομίζω ότι κατάλαβα από τα λόγια του Επιτρόπου Δεγούχτ. Και από τα λόγια των προαλυσάντων. Τι αρμοδιότητε που βλέπουμε να μοιράζονται σήμερα οι δύο επίτροποι. Τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει ο Μέν και η Δε. Δεν θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε μια αντίφαση που υπάρχει. Ο τομέας της αλίας έχει ρόλο θεμελιώδη και οι αλίες. Δεν πρέπει να μειώνουμε τις δυνατότητες και το δυναμικό τους ως προς την απασχόληση. Ε, εδώ υπάρχουν απαιτήσει της θάλασσας. Αν δεν θέλουμε οι αλληλείς μας να καταψύχονται σε μια κατάσταση μηδενικής απασχόλησης στην Ευρώπη θα πρέπει να κάνουμε κάτι στην Ευρώπη. Η Επίτροπος Δαμανάκη, η επίτροπο Δεκούχτ, είπαν ότι θα αφοσιωθούν εξ ολοκλήρου στο στόχο αυτό. Όμως νομίζω ότι έχουν μια κοινή πολιτική γραμμή και η πτυχή τη Επιτρόπου Αλία με όλα όσα συμπεριλαμβάνει στις αρμοδιότητές του θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτή τη σημαντική προοπτική που θέτει η εκθεσή μα για το μέλλον. Ευχαριστώ, ευχαριστώ συνάδελφοι. Παρακαλώ όμω να περιορίσετε τον χρόνο σα, γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει. Ο κύριο Καπόλα Σάντου για του σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροποι, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, τα αλληλευτικά προϊόντα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργεια είναι μια σημαντικότατη συνιστόσα τη διατροφική αλυσίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω όλοι ξέρουμε. Και εμεί εισάγουμε 60% των αναγκών μα σε αυτή την κατανάλωση, όπω πολύ σωστά ανέφερε η Επίτροπό μα. Αυτό το απλό γεγονό αποδεικνύει την σημασία τη έκθεση του συναδέλφου Καντέκ. Και εγώ είχα την ικανοποίηση να συνεργαστώ μαζί του και ο για ένα θέμα τόσο σημαντικό και αναζητώντα τρόπου να, να, να περισπιστούμε αυτόν τον τομέα και την απασχόληση που συμπεριλαμβάνει και του Ευρωπαίου καταναλωτέ. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες λοιπόν συμφωνούν με τις συστάσεις και τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης και ιδιαίτερος με ό,τι αφορά τις συστάσεις και τις ανησυχίες που εκφράζονται ως προς την ανάγκη να διασφαλίσουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τα περιβαλλοντικά κριτήρια που πρέπει να ισχύουν για την εισαγωγή, την παραγωγή και τη μεταποίηση των ίδιων αυτών προϊόντων. Η έκθεση πολύ σωστά προσεγγίζει και άλλα θέματα που θα έπρεπε να υποστηρίξουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Και βεβαίω η ομάδα μα θα υπερψηφίσει την έκθεση αυτή. Και ευχαριστούμε τον συνάδελφο Κάντεκ για το εξαιρετικό του έργο. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριο Γκάλαγκερ για του ε, ελεύθερου δημοκράτε. Για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κυρία και κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστώ τον συνάδελφο Κάντεκ για την έκθεση αυτή η διαρκή κατρακύλα των τιμών της αλίας τα τελευταία χρόνια είναι αποτέλεσμα βέβαια άμεσο των μαζικών εισαγωγών αλληλευτικών προϊόντων έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εκεί δεν τηρούνται οι αυστηρές προδιαγραφές που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι υγειονομικές, ούτε οι προδιαγραφές αηφορίας. Έρχονται λοιπόν τα προϊόντα αυτά στην ευρωπαϊκή αγορά σε τιμές οι οποίες συνθλίβουν τους ευρωπαίους παραγωγούς. Στο πλαίσιο λοιπόν τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική, πρέπει το ζήτημα αυτό να αντιμετωπιστεί. Και γνωρίζω ότι η Επίτροπο κυρία Δαμανάκη θα το αναλάβει το θέμα αυτό και θα το αντιμετωπίσει. Γιατί Έχουμε να κάνουμε με πολύ σημαντικά προϊόντα, όπως είπαν και οι δύο επίτροπε, η πατρίδα, και οι δύο επίτροποι. Η πατρίδα μου κάνει εισαγωγές προϊόντων σε ύψος 181 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο καταναλωτής δεν είναι ενημερωμένος για την προέλευση των προϊόντων αυτών. Έτσι λοιπόν η υπαγωγή εξαγωγών θα πρέπει να στοχεύει στη μείωση του 66% σε 50% μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Για να το καταφέρουμε όμως αυτό πρέπει και να αποδιαρθρώσουμε τη γραφειοκρατία που επιβαραίνει τους παραγωγούς μας. Πρέπει να απλωστεύσουμε τις, τις γραφειοκρατίες, όλες οι γενικές διευθύνσεις και όλα τα αρμόδια ε, τμήματα των κρατικών μηχανισμών στα κράτη-μέλη πρέπει να ε, βοηθήσουν σε αυτό το στόχο. Η κυρία Λεβίν για 1,5 λεπτό και ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, κυρία και κύριε Επίτροπε, καλωσορίζω και εγώ την έκθεση ΚΑΝΤΕ για τις εισαγωγές ε, αλληλευτικών προϊόντων. Τα αλληλευτικά αποθέματα έχουν μειωθεί πολύ σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλο ποσοστό των ε, ψαριών που καταναλώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται από, την άλλη, από την, τις ε, εισαγωγές. Δεν θα ήταν όμως υποχρεωτικό κάτι τέτοιο εάν είχαμε μια συνεπή πολιτική για τα αλληλευτικά αποθέματα και τα ενισχύαμε έτσι ώστε να έχουμε αηφόρο αλία. Ούτε και χρειάζεται στη τελευταία ανάλυση να εξάγουμε τα δικά μας αλληλευτικά προϊόντα σε τρίτες χώρες. Υπάρχουν συμφωνίες που μπορεί να αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμφωνία IUU επί παραδείγματι, δηλαδή ε, την υποχρεωτική πιστοποίηση όλων των αλληλευτικών προϊόντων που μπαίνουν σε ευρωπαϊκές αγορές, που να δείχνουν, που, ε, που να δείχνουν τα πιστοποιητικά που και με ποιες συνθήκες έχουν ε, παραχθεί ή ε, πιαστεί τα ψάρια αυτά. Και επίσης ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι από ορισμένε χώρες, ιδιαίτερα τις ε, χώρες εκείνε του κόσμου, στις οποίες κρατεί η διαφθορά, είναι πολύ εύκολο τέτοια πιστοποιητικά να πλαστογραφηθούν, να ετοιμαστούν χωρίς καμιά δυσκολία. Πρέπει λοιπόν εμείς να έχουμε εκείνου τους πόρους που θα μας επιτρέψουν να πιέσουμε και να εξασφαλίσουμε τις ε, προδιαγραφές που θέλουμε. Επίσης υπάρχουν μέσα από τα Ηνωμένα Έθνη τα, τα οποία μέσα, την οποία νομοθεσία πρέπει όμως να εφαρμόσουμε όπως πρέπει. Το 2006 είχε εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα της, ε, ε, το, το ενδεχόμενο εφαρμογής των συνθήκων περί ευθύνης, υπεύθυνης αλίας της FAO. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κρομπάσικς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ καλή έκθεση των κύριο Καντέ. Είναι μια ισορροπημένη έκθεση που καλύπτει όλη την αλληλευτική πολιτική και την ε, εξέλιξη της μέσα από την αναθεώρηση. Βλέπουμε πώς είναι οι τομείς ε, της κοινή αλληλευτικής πολιτικής που διαφοροποιούνται ριζικά από αυτά, ε, των οποίων η κατάσταση μάλλον διαφοροποιείται ε, ριζικά από αυτά τα οποία ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από αυτά που μας λέτε. Και οι αλείς μας λένε όντως ότι πρόκειται και μια ύψιστη σημασίας έκθεση. Η αλλιευτική πολιτική πρέπει να την λάβει σοβαρά υπόψη της. Κύριε Επίτροπε, σε πολλές συναντήσεις μας ακούσαμε να λέτε ότι η κοινή αλληλευτική πολιτική πρέπει να αποκτήσει ένα νέο πρόσωπο, να, να διαμορφωθεί. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση αποτελεί την εναλλακτική για τις ε, ιδέες που θα σχηματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από την αναθεώρηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντούτζ έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπη, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους, ε, τον εισαγητή για την έκθεσή του και να πω ότι στις 24 Ιουλίου 2008 το... με την οικονομική κρίση που έπληκε τον ευρωπαϊκό αλληλευτικό στόλο, η, τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Μέλωση ενέκριναν προσωρινά μέτρα για την αναδιάρθρωση και αναστήσταση του στόλου. Πολλοί αλλοί προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν αυτά τα μέτρα, αλλά χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν και τι συνθήκε διεθνού οικονομική ύφεση. Η τιμή των ε, γαρίδων και των καραβίνων που πουλούνται στη Βόρεια Ιρλανδία ε, πλήγει ιδιαίτερω από τα μέτρα αυτά, ενώ οι εισαγωγέ οστρακοειδών είναι πλέον πολύ μεγαλύτερε. Χρειαζόμαστε βεβαίω ψάρια στην Ευρώπη, αλλιευτικά προϊόντα, αλλά να μην τα φέρνουμε με οποιοδήποτε κόστο μέσα από τα σύνορά μα. Θα πρέπει να δούμε και τις επιδοτήσεις προς τους αλλοίς και να δούμε τι γίνεται με τις αντιφάσεις αυτές που προκαλούν οι άρσεις των επιδοτήσεων και την ταυτόχρονη εισαγωγή αρρύθμιστων και μη ελεγμένων αλληλευτικών προϊόντων που υπονομεύουν την αηφορία και την διάρκεια ζωής που θέλουμε να πετύχουμε για την δική μας ευρωπαϊκή βιομηχανία. Εδώ λοιπόν υπάρχει έλλειψη συνέπειας. Θα πρέπει να αντιστρέψουμε αυτές τις τάσεις και αυτό στηρίζω την έκθεση του κυρίου Καντέκ. Σας ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, για όσους ήρθατε να ψηφίσετε, θα ψηφίσουμε στις 12 και 20. Εάν θέλετε λοιπόν μέχρι τότε να παραμένετε λίγο ήσυχοι για να ολοκληρώσουμε την έκθεση αυτή. Και τώρα η κυρία Φράγκα Στέβερ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Η έκθεση αυτή έρχεται επειδή το ζήτησε ουσιαστικά ο τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο λιευτικός τομέας, ο οποίος δεν ζητάει προστατευτισμό. Ζητάει όμως, εδώ που έχουμε φτάσει και δεδομένων των τάσεων που παρατηρούμε και των όσων μας λέει η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, ζητάμε την έκθεση του κυρίου Καντέκο στις διαπραγματεύσεις που γίνονται για τα κεφάλαια αλίας να βγουν από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και να πάνε στη Γενική Διεύθυνση Μάρε. Το ίδιο και για την υδατοκαλλιέργεια, γιατί μιλάμε για ιδιαίτερα ευαίσθητα προϊόντα. όπω για παράδειγμα ο τόνο. Και μια που μιλάμε για τόνο, το έχουμε το παράδειγμα στις συμφωνίες ε, με την Παπούα, Νέα Γουινέα και τα Φίτζι. Με τις παρεκκλήσεις που έχουμε από τον κανόνα για την προέλευση των προϊόντων, με αποτέλεσμα οι Ταϊλάνδοι και οι Φιλιππίνες ανταγωνιστές μας να μπορούν κάτω από πολύ καλύτερες συνθήκες να έχουν τον δικό τους ηλεκτρικό τομέα. Λοιπόν, χάρη στη δικιά σα την ε, πολιτική, η Παπούα έχει περισσότερες θέσεις απασχόλησης, ποιότητα. Το ξέρετε αυτό. Ξέρετε τις καταγγελίες που έχουν κάνει μη κυβερνητικέ οργανώσεις για την δουλειά ε, που γίνεται όμως από τα παιδιά που δουλεύουν στα εργοστάσια. Ξέρετε την ε, καταστροφή που γίνεται στο περιβάλλον από την παράνομη αλία. Δεν είναι δικιά σας ευθύνη να αποφύγετε τέτοιες καταστάσεις. Ευχαριστούμε κύριε Φράγα. Ε, ο κύριος Κάλεγκερ έχει διαδικαστικό. Μικρόφωνο παρακαλώ. Η κατάσταση των ευρωβουλευτών εδώ είναι απαράδεκτη. Σε κανένα άλλο κοινοβούλιο στον κόσμο δεν θα είχαμε μια τέτοια κατάσταση. Κανένα σεβασμό δεν δείχνουν ούτε στην πρόεδρο τη Επιτροπή Αλία, ούτε σε κανέναν άλλον. Να σταματήσει η συνεδρίαση, παρακαλώ, μέχρι να δείξουν οι ευρωβουλευτέ εδώ ότι σέβονται το σώμα. Κύριε Γκάλαγκερ, πρέπει να συνεχίσουμε. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι ότι θα ζητήσω από όλου του συναδέλφου, παρακαλώ, μην κάνετε πηγαδάκια, 10 λεπτά υπομονή ακόμα να τελειώσουμε με αυτή την τόσο σημαντική έκθεση και τόσο σημαντική δουλειά και μετά ψηφοφορία. Ο επόμενο ομιλητή, η επόμενη ομιλήτρια μάλλον, η κυρία Ρότερ. Αξιότιμε Πρόεδρε, Αξιότιμη κυρία Μαρία Δαρμανάκη, η ευρωπαϊκή αλλιευτική πολιτική αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Οι αλληλείς μας έχουν να αντιμετωπίσουν τα συρρυκνούμενα αποθέματα και ταυτόχρονα ένα άλλο και εντυνόμενο αθέμητο ανταγωνισμό. Πρέπει κατεπηγόντως να προχωρήσουμε σε ριζοσπαστικές, σε ριζικές μεταρρυθμίσεις για να διαφυλάξουμε την επιβίωση της Ευρωπαϊκής Αλίας. Συμφωνώ με την κυρία Δαμανάκη ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε με όλο και περισσότερες ε, απαιτήσει τους αλληλείς μας με μεταρρυθμίσεις οι οποίες τους πιέζουν ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνουμε την αγορά. Είναι υπερβολικό να, τους, να απαιτούμε τόσα πολλά από αυτούς. Ο ανταγωνισμός το μόνο που χρειάζεται ή αυτό που χρειάζεται καταρχάς είναι την ανάκτηση των αλλιευμάτων μας, των αποθεμάτων μας των αλλιευτικών. Και πρέπει να είναι και ο καταναλωτής διατεθειμένος να πληρώνει πιο ακριβά το ψάρι που θα φάει προκειμένου να διαφυλάξει και την επιβίωση, να διατηρήσει την ε, αλία μας στην Ευρώπη. Η κυρία Ράιμερς, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κυρία Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κάντεκ για την πολύ καλή, επιτυχημένη, ισορροπημένη έκθεσή του, για όλους τους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία Έχουμε μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας, στην και πολιτική. Η ευρωπαϊκή αγορά έχει 12 εκατομμύρια τόνους ε, όγκο και 55 δισεκατομμύρια ευρώ αξία. Είναι η μεγαλύτερη δηλαδή του κόσμου. Αναπτύσσεται ταχύτατα και εξαρτάται από τις εισαγωγές, από τρίτα κράτη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και απαραίτητο να είμαστε σε θέση τα προϊόντα αυτά τα οποία εισάγουμε, τα προϊόντα αυτά τα οποία έχουν παραχθεί σε τρίτα κράτη, να τα ελέγχουμε έχουμε, καταβάλει, έχουμε καταθέσει τροπολογία όπου διατυπώνουμε τις ανησυχίες μας για την ε, ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι από απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης, χωρίς βέβαια να μπορούμε να κατηγορούμε για τα πάντα την απελευθέρωση της αγοράς. Δεν μπορούμε να... Το χρόνο σας τελείωσε, λέει ο κύριος Πρόνος. Και κλείνει το μικρόφωνο. Με συγχωρείτε, αλλά είμαι υποχρεωμένο να σα διακόψω. Ο κύριο Βαλένσα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, δεν έχω χρόνο αρκετό για να μιλήσω, άρα θα υπογραμμίσω απλώς και μόνο αυτό που με ενδιαφέρει, το πιο σημαντικό δηλαδή, το σχετικό με την έκθεση του κυρίου Καντέ πρέπει την αλία να την αντιμετωπίσουμε όχι σαν κάθε κοινό προϊόν παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε και τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου περί ευαίσθητων προϊόντων. Και γι' αυτό ευχαριστώ τον κύριο Κάντε, ο οποίο εξήρε την ιδιαιτερότητα του προϊόντος αυτού, του αλλιεύματο. Είναι πολύ σημαντικό στα προϊόντα της αλίας ή δυνατόν να ε, επιβάλλουμε την ε, αναγνώριση της ιδιαιτερότητάς τους ως ευαίσθητων προϊόντων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τρότμαν για ένα λεπτό. Παρακαλώ κύριε Τρότμαν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον συναδελφό μας Καντέκ για την εξαίρετη δουλειά του. Το κείμενο που ψηφίζουμε σήμερα δείχνει μια εξέλιξη όσον αφορά τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ιδέα των ελεύθερων συναλλαγών. Δεν μιλάμε για προστατευτισμό, αλλά η γραμμή που στηρίζουμε εδώ είναι λιγότερο αφελής. Συμφωνούμε όλοι για το ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή δεν φτάνει. Αντί να προσφεύγουμε σε εισαγωγές, κατά πρώτο λόγο, καλύτερα θα κάνουμε να διατηρήσουμε τα δικά μας αποθέματα προσφεύγοντας ακόμα και στην υδατοκαλλιέργεια, έτσι ώστε να διατηρηθεί ο τομέας και οι θέσεις απασχόλησης αυτών και προκειμένου να έχουμε μια αλία λιγότερο εξαρτώμενη από το εξωτερικό. Τώρα, όσον αφορά τι εξαγωγέ, να ξέρουμε ότι η αγορά των προϊόντων αλία και υδατοκαλλιέργεια να μην έχει αθέμητο ανταγωνισμό εξαιτία συνθήκων κοινωνικών ή φυτογενομικών που δεν ελέγχονται. Γι' αυτό λοιπόν και είμαι υπέρ σύμφωνα με τις δικές μας προδιαγραφές, κοινωνικές και τεφετογενικές, να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σήμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Πατράου Νέβες για ένα λεπτό τώρα. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η ευρωπαϊκή αγορά των αλληλευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ε, 60% ε, εισάγει τα προϊόντα που καταναλώνει. Η ευρωπαϊκή λοιπόν η κοινοτική αγορά στο προσεχέ μέλλον δεν θα είναι επαρκή για να καλύπτει την ζήτηση αυτών του είδου προϊόντων. Διότι έτσι, και τελικά έτσι οι εισαγωγέ μα θα γίνουν επιβαλλόμενη ανάγκη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε δύο σημαντικέ πτυχέ. Πρώτα απ' όλα ότι χρειάζεται η δημιουργία των κατάλληλων προποθέσεων, των αναγκαίων προποθέσεων για να εξασφαλίσουμε στον κοινοτικό καταναλωτή πρόσβαση στα αλληλευτικά προϊόντα και προϊόντα υδατοκαλλιέργεια που εισάγονται αλλά που πρέπει να είναι ποιότητα. Έπειτα, την θέσπιση ενό πλαισίου ανταγωνισμού θεμητού νομίμου και για τα εισαγόμενα προϊόντα και για αυτά που παράγονται και αλλιεύονται από τον τομέα αλλίας και τα το καλλιέργεια της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα που εισάγουμε σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ίδιες περιβαλλοντικέ κοινωνικές και ε, ποιοτικές προδιαγραφές που επιβάλλονται και για την κοινοτική παραγωγή. Και επειδή θα αναδιαρθρώσουμε την κοινή οργάνωση αγορών των προϊόντων αλλία και υδατοκαλλιέργεια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη του μηχανισμού που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε να σταδιακά να περιοριστούν οι δασμοί και να φροντίσουμε την μετριασμένη αύξηση των εισαγωγών. Θα πρέπει λοιπόν να εγκριθεί η έκθεση του Κοινοβουλίου που είναι και επίκαιρη και εγκρίνει ένα σύνολο προτάσεων εύστοχων για την προστασία του τομέα της αλίας και όσων κλάδων συνδέονται με τον τομέα της αλίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συνάδελφοι, για άλλη μια φορά, θα σας παρακαλέσω και να δείξετε και να μείνετε σιωπηλοί. Έχουμε το διαδικασία κάτι στη με τρει ομιλητέ. Παρακαλώ λοιπόν παραμείνετε για λίγο ήσυχοι, για πέντε έστω λεπτά. Η κυρία Άντρες Μπαρέα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο Δαμανάκη, ευχαριστώ και τον Επίτροπο Μπορείου που βρίσκονται εδώ για μια έκθεση πολύ σημαντική, το καθεστώς εισαγωγής. Δεν πρόκειται να επαναλάβω εδώ όσα είπαν οι προηγούμενοι, θα είμαι σύντομη. Για το θέμα της Ελίας είναι πολύ σημαντικό και φαίνεται ότι έτσι κι εδώ πέρα η κίνηση είναι τεράστια μέσα σε αυτή την αίθουσα πριν ψηφίσουμε. Το βασικό τι είναι, είναι ότι δεν έχουμε αυτάρκεια, ότι υπάρχει τεράστιο ανταγωνισμό, μερικέ φορέ αθέμητο. Εμεί πρέπει να διασφαλίσουμε την Ευρωπαϊκή Αλία, να αποφύγουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Θέλω να απευθυνθώ εδώ στον Επίτροπο για το Εμπόριο. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η αλία σαν ένα προϊόν που δεν είναι ευαίσθητο. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους κανόνες. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα προϊόν σαν να είναι βιομηχανικό. Είναι ένα ευαίσθητο προϊόν. Και γι' αυτό πρέπει να μπει κάτω από τις προδιαγραφές ε, του ΠΟΕ και του ΦΑΟ. Θέλουμε αηφορία. Δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τα είδη. Δεν μπορούμε να φροντίσουμε να έχουμε καλή πρόσβαση στην αγορά αν δεν θεωρήσουμε την αλία ευαίσθητο προϊόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Όπως είπα και πριν, αφήνουμε τη διαδικασία Catch και θα δώσω το λόγο στους επιτρόπους ευθύ αμέσω. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ ησυχάστε λίγο, σας παρακαλώ. Όλοι θέλουμε να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι επίτροποι απαντώντας τις ερωτήσεις των ευρωβουλευτών μας. Ησυχάστε λοιπόν. Για διαδικαστικό κύριε Atkins. Πρόεδρε, και πάλι προτείνω μέσω ημών, με ύψιλον να πάτε στην διάσκεψη των Προέδρων και να τους πείτε ότι πρέπει να ε, κανονίσουν καλύτερα το πρόγραμμα. Κάθε πέντε λεφτά από τις 12 και μετά αλλάζει η ώρα των ψηφοφοριών. Έχουμε κάποιο αεροπλάνο να πάρουμε. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει κάποιος στο κοινοβούλιο. Κάποιος πρέπει να τους το εξηγήσει αυτό. Κοιτάξτε, είχαμε πει ότι αναβάλλονται για τις 12 και 20 ψηφοφορίες εξ αρχής. Λοιπόν, παρακαλώ, επιτρέψτε να προχωρήσουμε στις απαντήσεις των επιτρόπων και στις 12 και 20, βεβαιώ, θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Η Επίτροπος κυρία Δαμανάκη. Πρόεδρε, ευχαριστώ δεν μπορώ να κάνω το πρόγραμμα όπως θα θέλατε, αλλά προσπαθώ να είμαι σύντομη. Και θα ήθελα να δώσω απαντήσεις στις ερωτήσεις των κυρίων και κυριών βουλευτών. Είπαμε και ο κύριος Δεγκού και εγώ ότι προσπαθούμε να βρούμε μια λεπτή ισορροπία. Πρέπει να έχουμε και βιώσιμο κλάδο στην Αλία και να εκπληρώσουμε τι υποχρεώσει μα προ τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και λοιπά διεθνή σώματα. Και γι' αυτό σα διαβεβαιώ όλου ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμβάλλουμε στην στο στόχο μια κοινή αλλιευτική πολιτική, μια μεταρρύθμιση τη κοινή αλλιευτική πολιτική που θα είναι πράγματι προ όφελο των αλλιέων μα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο, την κυρία Δαμανάκη, και δίνω το λόγο, εάν τον επιθυμεί, στον εισηγητή κύριο Κάντε. Ναι, θα ήθελα να μιλήσω. Ναι, Πρόεδρε, το επιθυμώ. Καταρχάς, θεωρώ ότι η συμπεριφορά των συναδέλφων στερείται κάθε σεβασμού, είναι απαράδεκτη σε κοινοβούλιο όπως το δικό μας σώμα, μας ντροπιάζεται μας ντροπιάζετε, το μόνο που σας ενδιαφέρει να ψηφίσετε και να γυρίσετε στα σπίτια σας. Έχουμε να επεξεργαστούμε μια πολύ σημαντική έκθεση, να έχετε τουλάχιστον το σεβασμό να ακούσετε τον άλλον. Διαφορετικά σκοφτείτε φύγετε από εδώ μέσα. Και μια και τα έβγαλα τα νεύρα μου, κυρίε και κύριοι, επιτρέψτε μου να σα πω το εξή. Σε ένα-δύο λεπτά θα έρθετε να ψηφίσετε και παρακαλώ να ψηφίσετε συντριπτικά υπέρ τη έκθεση. Και μια και έχω την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στην Επιτροπή Ελληνίας και την κυρία Φράγα, την πρόεδρό μας, που δέχθηκαν να αναλυφθεί αυτή η έκθεση και την ανέθεσαν σε μένα. Επίσης ευχαριστώ τον κύριο Καπούλα Σάντος, την κυρία Ράιμερς, τον κύριο Πρόφη και την κυρία Λόβιν, τους σκιώδεις ηγητές για τη συμβολή τους σε κάθε συζήτηση και στην επεξεργασία τροπολογιών. Ιδιαίτερα θα ευχαριστώ και όλους όσοι προσέφεραν τροφή στην έκθεση αυτή, τους εργαζόμενους από τον τομέα που με βοήθησαν ιδιαίτερα τους υπαλλήλους της DigiTrade και της ε, DigiMare, ε, τη Μαρία Γκαρσία Φερέρ, της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, τον Πιέρ Άμιλα, τον Ραμπό και τον Χουάν Ρανκό της DigiMare. Και ευχαριστηρώ ιδιαίτερος εσένα αγαπητή μου Μαρία που είσαι εδώ σήμερα, καλώς και τον κύριο Ντεγκούχτ. Οι απαντήσει σα, κύριε Ντεγκιούχτ, δεν ήταν απαντήσει, βέβαια, διότι προηγήθηκαν των ε, δικών μου παρατηρήσεων, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν με ικανοποιούν. Ωστόσο, ευχαριστώ και του συναδέλφου ε, από την ομάδα μου και του βοηθού μου και ιδιαίτερο ιδιαίτερο μια αναφορά στον Φιλίπ Μπιστιά, ο οποίο με βοήθησε πολύ με την έκθεση αυτή και με παρακολούθησε στην σύνταξή τη. Με συνόδευσε και παρακαλώ για άλλη μια φορά να δώσετε την ψήφο σα στην έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Κατέκ. Κύριε Ντεγκούχτ, δεν απάντησε και δεν απάντησε επειδή είχε τεράστια φασαρία εδώ στην αίθουσα. Οπότε θέλω να ζητήσω συγγνώμη προς τους δύο επιτρόπους για τη φασαρία που επικρατεί στην αίθουσα. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες παρακαλώ.